Uh, uh, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, πρωτού υποδεχθούμε την κυρία Βίκη Φόρντ για την κοινή συνεδρίαση, θα ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις για την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Βάσει των χθεσινών αποφάσεων του, των συντονιστών, ο κύριος Βιέφκα ορίστηκε εισηγητής για την πρόταση οδηγίας για την ε, μεταρρύθμιση του πλαισίου για την ε, ε, του συστήματος αποζημίωσης και την τροποποίηση της, δια, της οδηγίας 2030. Επίσης, θα ζητηθεί εξοδότηση για ε, σύνταξη ε, γνωμοδότησης για την ε, τρισδιάστατη εκτύπωση όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Γιούρη, την ε, αστική ευθύνη. Τρίτον, συμφωνήθηκε να διοργανωθεί η κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για τα καταστατικά για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις στις 22 Μαρτίου του 2017. 4. Συμφωνήθηκε η Επιτροπή να ζητήσει εξοδότηση για πραγματοποίηση αποστολής στην Ισλανδία 22 με 24 Μαΐου και αποστολή στην Μολδαβία με ε, θέμα το δικαστικό σύστημα. 5. Η, η Επιτροπή θα υποβάλει προφορικό ερώτημα για την ε, ισορροπία των φύλων στο δικαστήριο και θα ζητηθεί εξουδότηση για την διοργάνωση δύο ακροάσεων το 2017, συγκεκριμένα για το σύστημα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τις ε, εξαιρέσεις σε αυτό το σύστημα και τις ε, εκπομπές διαδικτυακής τηλεόρασης. Αυτά ως προς τις ανακοινώσεις. Περιμένουμε ακόμη την κυρία Βίκη Φόρντ. Συγχωρείτε, είμαι κλεισμένος στο σανσέρ για πέντε λεπτά. Ε, χαιρετίζω όλα τα μέλη της ε, Γιούρη και της ΙΜΚΟ και την πρόεδρο της ΙΜΚΟ, την κυρία Βίκη Φόρτ, που δεν είναι πια στο σανσέρ. Στόχος της ακρόασης είναι να ακούσουμε τους συν εισηγητές και να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη και των δύο επιτροπών για τις τροπολογίες ε, που προτείνουν αυτοί οι δύο συνεισηγητές. Οπότε τώρα να δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στην κυρία Βίκη Φόρτ. Ναι, καλημέρα. Ευχαριστώ τους συνεισηγητές για αυτή την κοινή έκθεση. και τις ε, τροπολογίες με βάση ε, τις οποίες αποφασίσαμε να εγκρίνουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είπαμε ότι θέλουμε να συζητήσουμε και θέματα που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το πρώτο σχέδιο έκθεσης γιατί όλοι θέλουμε να δούμε τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μέσω τροπολογιών. Οπότε απευθείας να δώσω το λόγο στον κύριο Βος ο οποίος είναι εισηγητής της Τζούρι για να αλλάξουμε και επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε την κυρία Γκέπαντ και τους υπόλοιπους ε, σκιώδεις ή τους σκιώδεις. Νομίζω ότι έχουμε επιτύχει αρκετά για την προσέγγιση των απόψεών μας. Δεν έχουμε, δεν έχουμε συμπέσει απόλυτα, αλλά ήδη έχουμε προσεγγίσει η μεν τους δε. Αυτό που θέλουμε είναι νομική σαφήνεια για να αποφευθούν επικαλύψεις με άλλες νομικές πράξεις όπως η, ο βασικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων, η οδηγία για τους καταναλωτές, η επερχόμενη οδηγία για ε, τις Πρέπει λοιπόν να έχουμε και άλλα κείμενα, πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε τις διαφορές μεταξύ την, της οδηγίας για τα απτά αγαθά και για τα ψηφιακά αγαθά και πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό ο οποίος νομίζουμε αυτός ο διαχωρισμός θα πρέπει να είναι ανοιχτός προς το μέλλον αλλά τεχνικά ουδέτερος και ίσως λοιπόν να υπάρχει με αυτόν τον τρόπο νομική σαφήνεια και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις γιατί το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε για το θέμα αυτό είναι το λεγόμενο embedded software. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με λογισμικό θα πρέπει να υπάγεται στις αρμοδιότητες του ψηφιακού. Εκτός εάν ο πολιτής ή ο κατασκευαστής μπορεί να μας αποδείξει κάτι διαφορετικό. Επίσης επιχειρήσαμε και θα το επιχειρήσουμε ακόμη περισσότερο γιατί δεν το επιτύχαμε μέχρι στιγμή στην έκθεση να υπάρχει ίδια νομική αλληλουχία μεταξύ της οδηγίας των αγαθών και της οδηγίας για το ψηφιακό περιεχόμενο. να συμβαδίζουν όλα αυτά με την οδηγία για τους καταναλωτές. Αυτό που διευκρινίσαμε στο άρθρο 3 παράγραφος 8 είναι ότι ισχύει ε, ανεξάρτητα από την ε, οδηγία που εξετάζουμε τώρα ο βασικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων. Στο άρθρο 4α λέμε για να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια ότι οτιδήποτε είναι κατά του θεμελιώδους κανονισμού δεν ισχύει ή δεν είναι δεσμευτικό. Αυτό δεν θα πρέπει να ελεγχθεί λοιπόν ε, στο συμβατικό δίκαιο και θα πρέπει στο μέλλον να δούμε πώς μπορούμε να το διευκρινίσουμε περαιτέρω με μια αιτιολογική σκέψη. Δεν συμφωνήσαμε για τις ε, ε, προθεσμίες εγγύησης. Ίσως θα πρέπει να υπάρξει μια ιεράρχηση. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να επιδιώξουμε την πλήρη εναρμόνιση γιατί έτσι απλουστεύεται η κατάσταση και να επιτύχουμε και μια λογική ισορροπία με το επίπεδο προστασίας ε, του καταναλωτή και των δικαιωμάτων των παραγωγών και πολιτών. Για τα δεδομένα τώρα. Το εξετάσαμε πιο προσεκτικά. Ιδιαίτερα για τα προσωπικά δεδομένα, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Είπαμε λοιπόν ότι ο βασικός κανονισμός φυσικά πρέπει να ισχύει και για τα προσωπικά δεδομένα και όλα τα λοιπά στοιχεία πρέπει να διευκρινίσουμε ακόμη ακριβώς τι σημαίνει ακριβώς λοιπά στοιχεία και τι νομικές συνέπειες θα είχε αυτό. Για πρώτη φορά περιλαμβάνουμε αυτή την έννοια εδώ, αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται με την επιστροφή και την περαιτέρω χρήση αυτών των στοιχείων όταν θα λύγει το συμβόλαιο. Ένα περαιτέρω θέμα που θα είναι δύσκολο γιατί έχει να κάνει και με τον κώδικα για τις τηλεπικοινωνίες όπου τώρα αρχίζει να εκπονείται η νομοθεσία. Ένα θέμα λοιπόν είναι Τι θα αφήσουμε για να ρυθμιστεί από αυτό το κώδικα για τις τηλεπικοινωνίες, για παράδειγμα για τα κοινωνικά μέσα, τις υπηρεσίες μηνυμάτων. Τι θα πρέπει να περιλάβουμε λοιπόν στη δική μας οδηγία και τι ίσως είναι καλύτερα να ρυθμιστεί αλλού. Χρειάστηκε να ασχοληθούμε με πολλά θέματα. Το δικαίωμα για παράδειγμα ε, καταγγελίας ή προσωρινής διακοπής για μακροπρόθεσμα συμβόλαια και αυτό μας απασχόλησε και για την ε, ε, επιστροφή των δεδομένων εξετάζουμε όλες τις δυνατότητες. Ευχαριστώ. Η συνεισηγήτρια της ΙΜΚΟ για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την καλή συνεργασία που είχαμε κύριε Φως. Ευχαριστώ και τους σκιώδες γιατί οι συνεδριάσεις που έχουμε διοργανώσει από κοινού μας έχουν βοηθήσει πολύ και οδήγησαν στο να καταφέρουμε να επιλύσουμε ορισμένα τουλάχιστον από τα προβλήματα και αυτό είναι θετικό. Ένα από τα ερωτήματα με τα οποία ασχοληθήκαμε ήταν ο ορισμός του πεδίου εφαρμογής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα, διότι η πρόταση της Κομισιόν ήταν πολύ προβληματική ως προς αυτό, καθώς δεν υπήρχε μια σαφής οριοθέτηση μεταξύ αυτών που θα ρυθμίζονταν σε αυτήν την οδηγία και στην οδηγία για τα υλικά αγαθά. Το να ορίσει κανείς που υπάγονται τα δεδομένα, ε, σκέφτομαι για παράδειγμα τα, τα, τα smartphone πράγματι αφορούν μόνο τη, το, τα τηλεφωνήματα ή μήπως τελικά χρησιμοποιούνται όλο ένα και περισσότερο ως υπολογιστές. Γι' αυτό για νομική ασφάλεια είπαμε ότι όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τα δεδομένα θα πρέπει να υπάγονται στην οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο ε, και να ρυθμίζονται εκεί προκειμένου να μην, δημιουργούνται, να μην δημιουργείται αβεβαιότητα από νομικής άποψης και να αποσαφηνίζεται ακριβώς ποιο είναι το θέμα το οποίο αφορά η συγκεκριμένη οδηγία και γι' αυτό το λόγο ε, ε, χαίρομαι που η συνεργασία μου και με τον κύριο αριμό για την πρόταση για τα υλικά αγαθά είναι πάρα πολύ καλή γιατί και εκεί ε, δουλέψαμε τους ορισμούς προκειμένου να μην υπάρχουν κενά. Και αυτό είναι πολύ θετικό επίσης. Δεύτερο θέμα που μας απασχόλησε και είναι πολύ σημαντικό είναι πράγματι αυτή, αυτός ο τομέας της αντιπαροχής της πληρωμής με δεδομένα. Δεν το θέλουμε αυτό. Δεν μας αρέσει, ε, είναι, αλήθεια, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε την πραγματικότητα κατάματα και να παραδεχθούμε ότι αυτό συμβαίνει ήδη. Γι' αυτό ε, δεν γίνεται να πούμε ότι αυτό θα το παρακάμψουμε ή δεν θα το, θα το αφήσουμε εκτός της οδηγίας. Ε, υπήρξε και μια τέτοια ε, συζήτηση, γιατί αλλιώς τα πράγματα θα ε, ξεφύγουν από τον έλεγχο και είπαμε έτσι ότι θα ακολουθήσουμε την πρόταση της Κομισιόν αλλά θα προσπαθήσουμε να θεσπίσουμε σαφείς κανόνες προκειμένου να ε, ισχύει πλήρως και στο σύνολό του ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ε, και στο συμβατικό δίκαιο. Ε, εκεί λοιπόν καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες για να βρούμε την κατάλληλη διατύπωση αλλά νομίζω ότι καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι θετικό, είναι ε, κατάλληλο για, την, ε, για το συγκεκριμένο κείμενο. Σκέφτομαι και τα λοιπά δεδομένα. Είναι και μια καινούργια σχετικά συζήτηση. Ε, εγώ θα πρότεινα να μην κάνουμε τροποποιήσεις στην πρόταση της Κομισιόν γιατί υπάρχει την περίοδο αυτή μεγάλη αβεβαιότητα ως προς το μέχρι πού πηγαίνουν τα προσωπικά δεδομένα και είναι κάπως ασαφές αυτό το ζήτημα. Τα τα δεδομένα όπως έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή και το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στη Γερμανία ε, φαίνεται να επεκτείνονται όλο και περισσότερο αλλά ακόμη είναι ασαφές. Θα έλεγα λοιπόν να το ε, αφήσουμε στην πρόταση της Κομισιόν να μην ζητήσουμε την απαλήφή του για να ε, ενισχύσουμε αυτήν την νομική σαφήνεια που είναι απαραίτητη. Θα ήθελα επίσης να απαντήσω σε μια ερώτηση της κυρίας Ρέντα που δεν κατάφερα να την απαντήσω στην τελευταία ε, ε, συνεδρία των σκιωδών τη διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 12 ότι τα το ψηφιακό περιεχόμενο δεν μπορεί εύκολα να απεγκατασταθεί. Μιλούμε για δεδομένα που είναι για παράδειγμα αποθηκευμένα σε ένα USB stick. Προφανώς για εμάς τα δεδομένα αυτά ανήκουν στο ψηφιακό περιεχόμενο. Αν ε, υπάρχει ασάφεια ε, ε, μπορούμε να το ξαναδούμε για να το αποσαφηνίσουμε και να διασφαλίσουμε ότι αυτό ακριβώς αναφέρεται αλλά ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί άκυρες ρήτρε ε, για τα δεδομένα. Εκεί στο άρθρο 4 ε, ε, προσθέσαμε μία διάταξη ώστε αυτό να αναφέρεται και στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης για δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε για την αντιστροφή της, του βάρους απόδειξης, για τα δικαιώματα εγγύησης, για να σας αναφέρω κάποια από τα ζητήματα που εκκριμούν Εκεί θα χρειαστεί να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχουμε χρόνο για τους σκιώδεις ηγητές και των δύο να, να λάβουν το λόγο. Η κυρία Πάουνοβα είναι εδώ. Για δύο λεπτά παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Καλωσορίζω το σχέδιο της ε, έκθεσης ε, από τους δύο συνεισηγητές και τις προσπαθειές τους να βρουν ε, κοινό έδαφος για ορισμένα ζητήματα. Χαίρομαι που έχουν καταθέσει σαφείς προτάσεις. Υποστηρίζω τι λύσεις που δίνουν σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή και τους ορισμούς που θα μας βοηθούσαν να μην κατακαιρματίσουμε το κεκτημένο. Συμφωνώ επίσης με το ότι στο σχέδιο κειμένου γίνεται διάκριση μεταξύ των ορισμών του ψηφιακού περιεχομένου και των ψηφιακών υπηρεσιών. Νομίζω ότι με αυτό θα διασφαλίσουμε ε, μία στεγανή νομοθεσία για το μέλλον ε, και θα πρέπει ε, ουσιαστικά να έχουμε έναν ορισμό του ψηφιακού περιεχομένου και να συμπεριλαμβάνουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της πλατφόρμας, το iCloud, το υπολογιστικό νέφος και άλλους τέτοιους ορισμούς. Επίσης ε, βρέθηκε μια λύση για το ανθιτολογισμικό που πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι ένα θετικό βήμα προς το να πετύχουμε υψηλή προστασία των καταναλωτών. Εισάγοντας ένα σαφές κριτήριο σε σχέση με τα, ε, με τα αγαθά, τα ε, υλικά και το ψηφιακό περιεχομένο. Επίσης είδα και την έκθεση του κ. Χάρη για την για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε ευθυγράμμιση των δύο προτάσεων στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου να στοχεύσουμε σε περαιτέρω εναρμόνιση. Συμφωνώ και καλωσορίζω τις αποσαφηνήσεις ότι οι καταναλωτές μπορούν να σεβαστούν πλήρως στην προστασία υπό την GDPR και χαίρομαι συνένεση για αυτό το θέμα που αφορά και τους καταναλωτές, αλλά μειώνει και το άχθος για τις επιχειρήσεις, η εμπιστοσύνη στις ψηφιακές υπηρεσίες είναι σημαντική και είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των καινοτόμων υπηρεσιών στην Ευρώπη και προκειμένου να υλοποιηθεί και η ψηφιακή αγορά σε ό,τι αφορά την ανάκτηση των δεδομένων. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν έχει νόημα να κάνουμε ανάκτηση των δεδομένων σε όλες τις περιπτώσεις και αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν τα δεδομένα, όταν επιστρέφονται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις καταναλωτές. Περνήτως χάρη τα avatar σε παιχνίδια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, σε άλλα παιχνίδια, αλλά και τα νόημα δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και να κλείσω λέγοντας ότι είναι προφανές ότι οι δύο εισηγητές δεν έθιξαν μια σειρά πτυχών όπως το βάρος της απόδειξης, τα ένδικα μέσα, η καταγγελία μακροπρόθεσμων συμβάσεων και αυτό δίνει και χώρο στους κοιόδης εισηγητές να καταθέσουν περαιτέρω τροπολογίες για την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Ροζιέρα που σιάζει, ούτε ο κύριος Ντάλτον έχει έρθει ακόμη, ούτε ο κύριος Τζεμπάσκι. Oh, Ξέρω ότι έρχεται ο κύριος Ντάλτον, αλλά μου είπε ότι θα καθυστερήσει. Ας καθίσει η κυρία Ροζιέρ. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Κάλλας, να πάρει το λόγο δύο λεπτά, ο κύριος Κάλλας δεν είναι εδώ, αλλά εγώ μπορώ να πάρω το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ε, εισηγητές για την έκθεση αυτή θα ήθελα να τονίσω ένα σημαντικό σημείο. Εισαγαγούμε νέους κανόνες σε ένα τομέα σχετικά καινούριο και που μεταβάλλεται πολύ γρήγορα. Για πρώτη φορά συζητούμε αυτούς τους κανόνες και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε σαφήνεια δικαίου Επίσης, ασκούμε κριτική στα διάφορα επίπεδα ε, του δικαίου, του συμβατικού. Έτσι, λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ στο πώς διασυνδέονται οι διάφορες νομοθεσίες, κυρίως το GDPR ε, και η οδηγία σε ό,τι αφορά τις ε, αθέμητους όρους των συμβάσεων. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες αποσαφηνήσεις. Η αλλαγή στην, στο νόημα του εφοδιασμού ή ο ορισμός του λογισμικού περιεχομένου ή των υπηρεσιών και για τη διάκριση που γίνεται από τους εισηγητές μεταξύ του ψηφιακού περιεχομένου και των ψηφιακών υπηρεσιών, καλωσορίζω την προσέγγιση αυτή, δεδομένου ότι η προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου διαφέρει από τις ψηφιακέ υπηρεσίες και οδηγεί σε διαφορετική συμπεριφορά από τους καταναλωτές. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται διάκριση αν δεν γίνεται κάποια διαφοροποίηση στην έκθεση σε σχέση με αυτά τα δύο ζητήματα. Η ίδια συζήτηση έχει να κάνει με τις ελεύθερες υπηρεσίες. Είναι οι προσδοκίες των καταναλωτών, διαφέρουν. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα νόμο που να θέτει στο ίδιο επίπεδο το περιεχόμενο, το δωρεάν ή το επιπληρωμή. Γιατί να πληρώσει ο καταναλωτή για οτιδήποτε αν έχει τα ίδια δικαιώματα και μπορεί να έχει ελεύθερες ε, υπηρεσίες ε, ή δίνοντας προσωπικά δεδομένα για την τροποποίηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στον ψηφιακό κόσμο οι επικαιροποίησεις να γίνονται συνεχώς. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να διορθωθεί οποιαδήποτε ευαλωτότητα στο λογισμικό για να προστατευτούμε ε, και προκειμένου να έχουμε αυστηρούς, κάνοντας αυστηρούς το κανόνες τελικά μπορεί να βλάψουμε τους καταναλωτές παρά να τους προστατεύσουμε. Συμφωνώ για τον κύριο Βος, ε, για τα άλλα δεδομένα που πρέπει να αποσαφινιστούν. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για παραδείγματα όπως οι εικόνες και εκεί μιλάμε για περιεχόμενο που δημιουργείται από το χρήστη και όχι για δεδομένα. Αυτά ήθελα να πω εγώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ροζιέρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τους δύο συνεισηγητές γιατί μιλάμε για ένα θέμα ε, το οποίο ουσιαστικά είναι καινούριο, πρόκειται για μια πολύ σημαντική δουλειά και μιλάμε για την προστασία των καταναλωτών για αυτά τα προϊόντα. Έχουμε κάνει πραγματικά πρόοδους για τον Ευρωπαίο καταναλωτή, ιδίω ό,τι αφορά τον ορισμό του πεδίου εφαρμογή, που σε αυτό το στάδιο μας επιτρέπει να έχουμε έχουμε ε, ουσιαστικά επιμερισμό μεταξύ των δύο οδηγιών για την προμήθεια περιφερειακού χωμένου και για τα αγαθά, κυρίως όταν συμπεριλαμβάνουμε τα αγαθά τα οποία έχουν ένθετο λογισμικό και στην περίπτωση αυτή ε, αντιστρέφουμε το βάρος της απόδειξης ε, σε ό,τι αφορά την προέλευση και βλέπουμε τι γίνεται όταν είναι προεγκαταστημένο το λογισμικό στο αγαθό, όταν είναι ε, ουσιαστικά πλήρες μέρο του λογισμικού ή όταν δεν έχει εγκατασταθεί. Τότε εκεί θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι αποδείξεις σχετικά με την προέλευση και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική πρόοδος αυτή. Επίσης γίνονται κάποιες διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις ε, Είχαμε μια αρχική διατύπωση της Κομισιόν που ήταν αρκετά ασαφής και έπρεπε να αποσαφινιστεί. Και εδώ έχουμε τα πρώτα στοιχεία που μας επιτρέπει να δούμε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Επίσης, ε, θεωρώ ότι έχουμε μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση για τα κριτήρια συμμόρφωσης. Έχουμε για πρώτη φορά υποχρέωση συμμόρφωσης για το ψηφιακό περιεχόμενο. Και εδώ ήταν αμφισβητούμενη η πρόταση της Κομισιόν γιατί αυτή τη συμμόρφωση την εξαρτούσε από τη σύμβαση, δηλαδή ανάλογα με τις διατάξεις στην οδηγία και ευτυχώς το σχέδιο της έκθεσης προτείνει να επανέλθουμε σε ένα μοντέλο που έχει εγκριθεί παγκοσμίω ε, σύμφωνα ε, με ε, την συμμόρφωση ενός στόχου, έτσι όπως έχουμε στην οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Επίσης, διερευνούμε το θέμα της δυνατότητας καταγγελίας ε, της σύμβασης, κυρίως όταν υπάρχει τροποποίηση του ψηφιακού περιεχομένου και επίσης να δούμε και πώς συνδέεται με τον κανονισμό της προστασίας των δεδομένων που επιτρέπει οποιαδήποτε στιγμή να αποσύρει τα δεδομένα του καταναλωτή. Σας ευχαριστώ. Ζαν Μαρή Καβαντά. Όχι, όχι, δεν θέλω να χρονοτριβήσουμε άλλο. Είναι πολύ καλή αυτή η εργασία και αποτελεί πρόοδο. Ευχαριστώ τους δύο συνεισηγητές αλλά και τους άλλους. Ε, νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί τους και εκτιμώ πολύ την εργασία τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντόλσον. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που καθυστέρησα. Κυκλοφορία είναι ζώρικη στις Βρυξέλλες. Η άποψη της ομάδας μου και των μελών της ΙΜΚΟ έχουμε ανησυχίες ότι θα δημιουργήσει δυσχέρειες και κόστος για τις εταιρείες η εφαρμογή αυτή της οδηγίας. Μερικά συγκεκριμένα σημεία. Το επιχείρημα για τα επιχειρήματα, για τα δεδομένα. Και με ανησυχεί το ότι παραμένει αυτή η έννοια, δεν ξέρω τι επιδιώκει να επιλύσει. Δεν δέχομαι ότι το να πληρώνει κανείς για περιεχόμενο με προσωπικά δεδομένα δεν είναι το ίδιο με το να πληρώνει με χρήματα. Κανένα δεν θα να μου πει ότι ανησυχεί από του εκλογεί μου ότι τα δεδομένα του ε, αξιοποιούνται με τρόπο που του δημιουργούν δυσχέρε. Κανεί δεν μου είπε ότι αυτό θα πρέπει να περιληφθεί στην νομοθεσία, αλλά κυρίω από τη στιγμή που εξισώνει κανεί τα δεδομένα με ε, κόστος αυτό σημαίνει ότι όλες οι ελεύθερες ε, apps πρέπει να έχουν ε, το ίδιο επίπεδο ε, προστασίας του καταναλωτή και προδιαγραφών με τις apps για τις οποίες πληρώνεις. Αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα και δεν θα βοηθήσει την ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Και ξέρω ότι πολλοί καταναλωτές θα διαμαρτύρονται αν δεν θα υπάρχουν πια δωρεάν εφαρμογές. Για τα λοιπά στοιχεία. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα φυσικά πρέπει να επιστρέφονται μετά τη λήξη του συμβολέου. Αυτό νομίζω ότι είναι σαφές και το στηρίζω. Αλλά αν το επεκτείνουμε και στα λοιπά στοιχεία, θα έχουμε διάφορα προβλήματα. Πρώτον, ποια είναι αυτά τα λοιπά στοιχεία. Για παράδειγμα, σε ένα παιχνίδι ένα κάστρο που έχτισες στο παιχνίδι. Είναι και αυτό λοιπόν στοιχείο. Όταν ε, λήξει το συμβόλαιο θα πρέπει να σου δώσει πίσω η εταιρεία το κάστρο. Θα το δώσουν υπομορφή κωδικού που είναι άχρηστο εκτός του συγκεκριμένου λογισμικού του παιχνιδιού. Γιατί υπάρχουν τα πνευματικά δικαιώματα. Και δεύτερον, νομίζω ότι είναι κατά του πνεύματος του γενικού κανονισμού που αφορά που την ανωνυμοποίηση των δομένων. Θα πρέπει να τα ε, κάνουμε και πάλι προσωπικά για να του τα στείλουμε πίσω αυτά. Προσβλέπω στην ε, περαιτέρω συζήτηση με τους δύο συγκητές, αλλά πρέπει να τα διευκρινίσουμε αυτά τα δύο σημεία, γιατί αλλιώ θα δημιουργήσουμε δυσχέρειες για τους προγραμματιστές να εκπονούν ελεύθερες apps. Πρόεδρος, οι δύο συζητητές θέλουν να σχολιάσουν τα σχόλια των ε, σκιωδών. Η κυρία Γκέπαρντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις ε, διευκρινήσεις. Να αναφερθώ σε δύο θέματα. Η κυρία Καλάς αναφέρθηκε στο θέμα των λοιπόν στοιχείων, των μη προσωπικών. Τι εννοούμε. Είπατε ε, οι εικόνες δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Εγώ τα θεωρώ προσωπικά και υπάρχουν ε, και δικαστήρια που συμφωνούν με αυτή την ερμηνεία. Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικές αντιλήψεις για το τι σημαίνει προσωπικά δεδομένα. Αν θέλουμε να τηρηθεί το επίπεδο προστασίας του γενικού κανονισμού, πρέπει να φροντίσουμε ούτως ώστε το θέμα αυτό να παραμείνει ανοιχτό για να μην υπάρχει νομική ασάφεια τι είναι προσωπικό και τι όχι. Χρειαζόμαστε νομική ασφάλεια. Πρέπει λοιπόν να παραμείνει. Για τον κύριο Ντόλτον, ίσως υπάρχει παρανόηση. Παρακαλώ διαβάστε τι ακριβώς γράψαμε. Δεν λέμε ότι απαγορεύεται να πληρώνει κανείς με στοιχεία. Ευχαριστώ θα το έκανα. Δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι πρέπει να φροντίσουμε ούτω ώστε οι καταναλωτέ, οι πολίτε να έχουν και να διατηρούν πλήρη δικαιώματα επί των δεδομένων τους. Και αν γίνεται περαιτέρω επεξεργασία τους για τις υπηρεσίες, ας πούμε, είναι αναγκαίο αυτό, τότε πρέπει να υπάρχει η ε, ενημερωμένη συνένεση του καταναλωτή. Αυτό λέμε. Και είναι το, το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε, γιατί τα στοιχεία συλλέγονται, και επεξεργάζονται για διαφήμιση και για άλλα. Ένα πολίτη πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πει όχι. Δεν θέλω να λαμβάνω εξατομικευμένη διαφήμιση. Πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να εναπόκειται στους καταναλωτές αυτή η δυνατότητα και αυτό επιδιώκουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φως, τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω την αίσθηση ότι το θέμα των δεδομένων θα πρέπει να το εξετάσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια προκειμένου να υπάρξει μια κοινή αντίληψη. Ε, είναι σαφές, δωρεάν εφαρμογές θα συνεχίσουν να υπάρχουν και όταν πληρώνει κανείς με δεδομένα του, τότε εκεί, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο γενικός κανονισμός είναι σαφής για το ποια θα πρέπει να είναι η μεταχείριση αυτών των δεδομένων. Δεν δημιουργούμε ούτε νέα δικαιώματα, ούτε νέες ε, ιδέες, νέα σκεπτικά. Όχι. Ε, από, με βάση δηλαδή το ε, συμβατικό δίκαιο. Όχι. Θα ισχύει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Το έχουμε αποσαφηνίσει αυτό. Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται και ότι δεν θα υπάρχουν επικαλύψεις, γιατί τα προσωπικά δεδομένα έτσι και αλλιώς ε, τίθενται σε επεξεργασία και χειρισμό με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού. Δεν χρειάζεται να ε, θεσπίσουμε νέους κανόνες. Στα άλλα ζητήματα και στις, στα άλλα στοιχεία... Ε, Πράγματι πρέπει να το δούμε. Το είπε και ο κύριος Ντάλτον και η κυρία Κάλλας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεδομένων πραγματικά δεν έχει νόημα να υπάρξει επιστροφή των δεδομένων αυτών γιατί έχουν ανωνυμοποιηθεί ε, ή ψευδονυμοποιηθεί. Ε, εκεί πραγματικά θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα τι ε, επιπτώσεις θα έχει μια τέτοια διάταξη, γιατί αν υπάρχει υποχρέωση ε, να, ε, να, καθίστανται επαναταυτοποιήσιμα τα δεδομένα, εκεί πράγματι υπάρχει μια παραβίαση του γενικού κανονισμού, γιατί θα πρέπει κανείς να ξανα... Ε, προσδιορίσει, ταυτοποιήσει τα δεδομένα για να μπορεί να τα επιστρέψει. Θα πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις. Αυτό που ε, είναι σημαντικό είναι να υπάρχει ενημέρωση και διαφάνεια και βεβαίως ε, δικαίωμα ε, υπαναχώρησης, ανάκλησης, αλλά ιδίως σε αυτό που ανέφερε η κυρία Κάλλας, είναι, είναι πράγματι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε ε, βήμα προς βήμα για να αποφύγουμε τυχόν ε, επικαλύψεις που θα ήταν και εντελώς περιτές. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα και θα τα συζητήσουμε βεβαίως. Ε, επί της ουσίας όλοι θέλουμε μια καλή ισορροπία και μια ενδεδειγμένη ε, χρήση και χειρισμό των δεδομένων. Ε, θα δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να εντάξουμε αυτήν την ε, λογική, αυτό το σκεπτικό στο νομικό κείμενο. Κάποιους ομιλητές στο δικό μου κατάλογο είναι οι ε, σκεδείς εισηγητές ε, από την άλλη επιτροπή, Ντένις Δεγιό, Κογιον Μαστάλκα, Μαρκο Τζούλιο, Λάουρα Φεράρα, Τζούλια Ρέντα. Κάποιοι είναι εδώ στην αίθουσα και κάποιοι απουσιάζουν. Δεν βλέπω τον Ντένις. Γιώργη Μαστάλκα, ούτε, Τζούλια Ρέντα. Ευχαριστώ. Καταρχήν πιστεύω ότι η έκθεση οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήδη επιλύει κάποια σημαντικά ζητήματα. Κυρίως ε, πιστεύουμε ότι έχουν εισαχθεί κριτήρια για την ε, αντικειμενική συμμόρφωση. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κριτήρια και μην ε, αφήνουμε να ρυθμίζεται αυτό το θέμα από την τελική συμφωνία με το χρήστη Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προσδοκίες του καταναλωτή και το τι υποτίθεται ότι θα πετύχει αυτό το περιεχόμενο. Επίση, το θέμα των κεκτημένων των ένδικων μέσων είναι πολύ σημαντικό, κυρίω αν μιλάμε για μικρέ αγορέ MP3 για 99 λεπτά του ευρώ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν το θέμα των προσφυγών και ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογή, ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο προτάσεων είναι καλός θα πρέπει να δούμε τον ορισμό του ένθετου λογισμικού, του ένθετου περιεχομένου, ιδίως γιατί από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει μια συμφωνία ότι και το περιεχόμενο που δίνεται σε ένα μέσο ε, το οποίο ε, είναι ένθετο σε αυτό το μέσο θα πρέπει να καλύπτεται από την πρόταση. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία έχω αναφέρει στο έγγραφο εργασία και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα στο σχέδιο τη έκθεση. Θα καταθέσουμε τροπολογίε, όπω παραδείγματο χάρη θέματα όπω τα πολλαπλά κατεβάσματα για τα προσωπικά δεδομένα. Πιστεύουμε ότι έχουμε καλά στοιχεία στην γνωμοδότηση της ΛΥΜΠΕ μπορούμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να τα συμπεριλάβουμε για να λύσουμε τα θέματα της αλληλεπίδρασης με τον κανονισμό της προστασίας των δεδομένων και σε ό,τι αφορά τώρα την αντιπαροχή. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μπορούμε να φανταστούμε ότι υποβάλλουν δεδομένα ή περιεχόμενο ε, οι χρήστες. Και δεν θα περιγραφεί απαραίτητα ως προσωπικά δεδομένα το περιεχόμενο αυτό και νομίζω ότι κάπως πρέπει να το καλύψουμε αυτό στην πρόταση για τα λοιπά δεδομένα, any other data. Ίσως ε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε. Εγώ είμαι σκιώδης και για τις δύο επιτροπές, θα προσπαθήσω λοιπόν να μην ακρηγορήσω. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα χρήσης των δεδομένων αυτών ε, θα πρέπει ε, ουσιαστικά να επιστρεφούν όταν λήξει η σύμβαση και σε ό,τι αφορά τις ε, ζημίες. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και όταν μιλάμε για αυτές τις ελεύθερες εφαρμογές ε, όταν ε, παραδείγματο χάρη βάζει ε, κάποιος χρήστης να, μια εφαρμογή να χρησιμοποιηθεί δωρεάν από τους υπόλοιπους τότε εκεί δεν θα πρέπει να έχουμε θέμα ζημιών Επίσης, πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ της προμήθειας και της διάθεσης. Μπορεί να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Πότε, παραδείγματος χάρη, γίνεται προμήθεια μιας υπηρεσίας ή διατίθεται και υπάρχει και μια σειρά άλλων θεμάτων. Νομίζω πρέπει να δώσουμε μια προσοχή σε ό,τι αφορά τις άρνησης ε, επαρκής υπηρεσιών. Πρέπει να διασφαλίσουμε πώς η ασφάλεια λαμβάνεται υπόψη στους προμηθευτές και πώς επικαιροποιούνται οι συσκευές. Μίλησατε για δύο επιτροπές, γι' αυτό σε επέτρεψα να έχετε τόσο χρόνο. άρχισαμε να σημειώνουμε και τους υπόλοιπους που θέλουν το λόγο και παρακαλώ αν θέλετε να προσταθείτε στον κατάλογο, κάντε μας ένα νόημα. Ο κύριος Τσούλο. Είναι εδώ η κυρία Φεράρα. Όχι. Θα ήθελε κάποιος άλλος συνάδελφος το λόγο. Κύριε Στατημάιερ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, καλωσορίζει η Κομισιόν ε, τη συνεργασία των δύο εισηγητών. Έχει γίνει ήδη δουλειά εις βάθος. Και καλωσορίζουμε ότι η δουλειά και για την ε, επιγραμμική πώληση αγαθών προχωρά παράλληλα. Είναι μια πολύ χρήσιμη προσέγγιση. Θέλω να σχολιάσω ένα σημείο που ανέκυψε στα σχόλια σχόλια όλων των βουλευτών. Το θέμα της συμπερίληψης δεδομένων και των λοιπών δεδομένων, είναι other data. Καλωσορίζουμε ότι και οι δύο εισηγητές ε, διατηρούν αυτή τη συμπερίληψη των δεδομένων στο πεδίο εφαρμογή. Ε, αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα αυτής της πρότασης για οδηγία. Όμως είναι σημαντικό να διατηρήσουμε και τα λοιπά δεδομένα. Και έχουμε δύο λόγους. Και τα λοιπά δεδομένα μπορούν επίσης να παρακολουθούν προσωπικά δεδομένα. Παραδείγματος χάρη, σκεφτείτε ότι κάποιος συλλέγει δεδομένα και, παραδείγματο χάρη, οι χρήστες ε, παρακολουθούν ε, μια συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά ε, για πόσο καιρό και ποιες είναι οι ηλικίε τους. Συλλέγονται αυτά τα δεδομένα χωρίς να συνδέονται με το άτομο που προσφέρει αυτά τα δεδομένα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χρήμα και να δοθούν σε κάποιον άλλο που θέλει να δημιουργήσει μια παρόμοια σειρά. Και αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χρήμα, αυτοί οι καταναλωτές έχουν λιγότερα δικαιώματα γιατί δεν συνδέονται τα δεδομένα πίσω με αυτούς. Διαφορετικά θα είχαμε μια αντίφαση με την GDPR, γιατί μία από τις κύριες αρχές είναι η ελαχιστοποίηση της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να αναγκάσουμε τους εμπορούς να ζητούν προσωπικά δεδομένα. Δεν έχει νόημα. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τα λοιπά δεδομένα στην πρόταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κάποια άλλα σημεία που σχετίζονται με την έκθεση των δύο συνσηγητών. Έχει, υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με τον ορισμό του φαδιασμού. Τη προμήθεια. λέει, ε, χωρίς την καθυστέρηση, αλλά όχι αργότερα από 30 μέρε. Αυτή προέρχεται από την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Κατανοώ ότι υπάρχει αναγκαιότητα εδώ να είμαστε συνεπεί με την ε, οδηγία περί καταναλωτών, όμω είναι πολύ σημαντικά να δούμε τι έγινε ε, σε ένα ανάλογο πλαίσιο, το ψηφιακό περιεχόμενο. Δεν έχουμε κόστο μεταφορά Στην άλλη οδηγία έπρεπε να ληφθεί υπόψη το κόστο μεταφορά. Τότε λέμε λέμε «Α, όχι αργότερα από 30 μέρες», τότε η πρακτική θα γίνει 30 μέρες και θα ζημιωθεί ο καταναλωτή. Δεν θα γίνουν νωρίτερα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, ε, εμείς ε, θα θέλαμε να μην γίνει αυτό για να μην ζημιωθεί ο καταναλωτή. Κάτι άλλο για το άρθρο 4α που αναφέρθηκε μερικέ φορέ. η σχέση του τέλου, αν ε, παραδείγματο χάρη ένα όρο τη σύμβαση παραβιάζει την οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα, εμείς Βλέπουμε ποιε είναι οι ανησυχίε των συγητών, ε, όμως τώρα ε, δεν αρμονίζεται στην GDPR και υπάρχει λόγος γιατί περιλαμβάνεται σε όλα τα κράτη ρήτρα ότι η αθέμητη όρη της συμβάσεις δεν είναι δεσμευτική. Έτσι λοιπόν, αν το βάλετε έτσι, οι έξυπνοι δικηγόροι θα σας πούνε «Α, τι σημαίνει, υπάρχουν κάποιο ε, λόγο που μπορεί να είναι, το χάρη, Παράνομε ρήτρε και δεν θα πρέπει να, να λαμβάνονται υπόψη. Έχω και άλλα σημεία, αλλά δεν προλαβαίνω σα τα πω. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ όλου του ομιλητέ και του εισηγητέ. Πραγματικά πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ακόμη, κυρίω για το θέμα των λοιπόν δεδομένων και να διασφαλίσουμε ότι είναι σαφή τα πράγματα και δεν έρχεται σε σύγκρουση με την ε, Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα και μου υπενθύμησαν ότι είχαμε μία κρόαση για παρόμοια ζητήματα ε, για, τα μακροπρό... για τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις. Είχαμε σκεφτεί να υπάρχει η δυνατότητα για νωρίτερο η καταγγελία της σύμβασης. Ίσως λοιπόν αυτές είναι κάποιες προτάσεις και για την επόμενη ε, φορά θα συνεχιστεί η συνεδρίαση της ΙΜΚΟ στο PHS 4.1. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συμμετοχή σας εδώ.